μετά από διαβούλευση των πολιτικών ομάδων το γεγονός ότι ο πρόεδρος προτείνει να αντιστραφούν τα δύο επόμενα ε, τα, τα εξή μάλλον σημεία στην ημερησία διάταξη και ζητώ την προσοχή σα. Το σημείο για την ασταθή κατάσταση στη Λιβύη και τι συνέπειε αυτού που αυτή τη στιγμή προβλέπεται για την Πέμπτη το πρωί θα εξεταστεί την Τετάρτη απόγευμα. Ενώ το σημείο που αφορά την 28η Σύνοδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον ΟΗΕ θα συζητηθεί την Πέμπτη το πρωί, ενώ τώρα προβλέπεται για την Τετάρτη το απόγευμα. Ε, έχετε αντιρρήσει, όχι. Οπότε τροποποιούμε την